Η ψηφοφορία θα γίνει στις 11.30 το πρωί της Πέμπτης. Προχωρούμε στο επόμενο θέμα, στην ημέρηση διάταξη. Πρόκειται για την ενδιάμεση έκθεση της κυρίας Χιούμπνα σε σχέση με την ε, χρηματοδοτική ενίσχυση χωρών των οποίων το νόμισμα δεν είναι το ευρώ. Και θέλω να ζητήσω από την κυρία Χιούμπνερ να λάβει το λόγο τέσσερα λεπτά. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. <clears throat> Η εστίαση για τις μεταρρυθμίσεις ε, με, λόγω της οικονομικής κρίσης ήταν κυρίως η, ευρωπαϊκή, ζώνη του ευρώ γιατί ήταν απαραίτητο να τροποποιηθεί η αρχιτεκτονική του ενίου νομίσματος. Καθώς προχωρούμε όμως στις μεταρρυθμίσεις δεν θα πρέπει να λησμονήσουμε την ανάγκη να διατηρήσουμε τη συνοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να διατηρήσουμε την ενότητα της ενιαίας αγοράς. Με τον τρόπο αυτό είναι απαραίτητο να υποστηρίξω ότι η μεταρρύθμιση της διευκόλυνσης για τις ε, ε, ενιαίες πληρωμές μπορεί να βοηθήσει χώρες που δεν είναι στη ζώνη του ευρώ και αντιμετωπίζουν μακροοικονομικές δυσκολίες. Είναι μια προσπάθεια να βοηθήσουμε τη διαδικασία για να πλησιάσουν οι χώρες αυτές με την ενίσχυση στο ισοζύγιο πληρωμών και μπορούν έτσι να εξασφαλίσουν ότι έχουν γραμμές χρηματοδότησης μέσα σε κατάλληλες συνθήκε. Έτσι θα μπορέσουν να αντιμετωπιστούν οι κίνδυνοι εγκαίρως και πρώιμα προτού γίνουν πραγματικές απειλές στην χρηματοπιστωτική σταθερότητα. Γιατί η κρίση και η εμπειρία της έδειξαν ότι μπορούν αυτές μετά να μεταδοθούν και να επιμολύνουν πολύ γρήγορα. Δεν δίδονται περαιτέρω δικαιώματα <clears throat> μόνο για περαιτέρω ε, βοήθεια, αλλά θεσπίζεται και μια σειρά από υποχρεώσεις όπως είναι τα μέτρα επιτήρησης και εποπτείας πριν και μετά από την παροχή βοήθειας. Οι κατευθυντήριες ε, γραμμές περιλαμβάνουν και προγράμματα μακροοικονομικής προσαρμογής επί τη βάση μιας ανάλυσης της βιωσιμότητας των δημοσίων οικονομικών. Με τον τρόπο αυτό μπορούμε να προωθήσουμε και ένα καλύτερο διάλογο σε διαθεσμικό επίπεδο σε σχέση με την χρηματοδοτική αυτή υποστήριξη της, ε, του ισοζυγίου πληρωμών. Θα πρέπει να ληφθεί επίσης και το δίπτυχο, το 2 που συνδυάζεται με τα θέματα της ε, χρηματοδοτικής υποστήριξης για τη ζώνη του ευρώ και έτσι θα αποτελέσουμε τμήματα μιας προσπάθειας εναρμόνισης για την ενιαία αγορά αυτή η ενισχυμένη υποστήριξη στο ισοζύγιο πληρωμών είναι πάρα πολύ σημαντική, ιδίω στο πλαίσιο τη Ευρωπαϊκή Τραπεζική Ένωση. Για να επιτύχει αυτή η Ένωση, τα μέλη τη θα πρέπει να αντιμετωπίζονται με ένα ισοδίκαιο τρόπο. Γι' αυτό τα μέλη που δεν είναι ακόμα στη ζώνη του ευρώ, που θέλουν να ενταχθούν στον ενιαίο μηχανισμό επιτήρηση, εποπτείες μάλλον, θα πρέπει να έχουν ένα κατάλληλο σύνολο από καθήκοντα και δικαιώματα. Ο στόχος αυτής της Ρύθμιση είναι να δοθεί μια δημοσιονομική εξασφάλιση για τις χώρες που δεν είναι στη ζώνη του ευρώ, γιατί οι αποφάσεις του ενιαίου εποπτικού μηχανισμού μπορούν να έχουν αρνητικές συνέπειες για όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ανάγκη για περαιτέρω ανακεφαλαιοποίηση. Από τη στιγμή λοιπόν που θα λειτουργήσει ο ενιαίος αυτός εποπτικός μηχανισμός, θα υπάρχει δυνατότητα της άμεσης ανακεφαλαιοποίηση όλων των τραπεζών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πιστεύω ότι η πρόταση αυτή θα πρέπει να περιλαμβάνει και ένα εργαλείο έμεσης ανακεφαλαιοποίησης για τις ε, τράπεζες των χωρών που συμμετέχουν στον ενιαίο εποπτικό μηχανισμό. Έτσι, θα μπορούν οι τράπεζες αυτές και οι κυβερνήσεις αυτών των χωρών να παίρνουν δάνεια για να μπορέσουν να ανακεφαλαιοποιήσουν τα πιστοτικά τους ιδρύματα. Ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθεροποίησης θα πάψει επειδή υπάρχει αυτός ο μηχανισμός, οι διευκόλυνση για το ισοζύγιο πληρωμών θα σταματήσει να ισχύει. Εν καιρό, αν υπάρξει μεταρρύθμιση της συνθήκης για τον ενίο μηχανισμό σταθερότητας, μπορεί να υπάρξει δυνατότητα να συμμετέχουν οι χώρες που δεν είναι στη ζώνη του ευρώ και συμμετέχουν στον ενίο εποπτικό μηχανισμό να συμβάλλουν στο μηχανισμό και στη χρηματοδότηση της ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών. Εν κατακλείδη, η μεταρρύθμιση του μηχανισμού υποστήριξη των πληρωμών δίδει μηνύματα τα οποία ξεπερνούν την χρηματοδοτική υποστήριξη και οδηγεί σε περαιτέρω εναρμόνιση των μεταρρυθμίσεων σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, που είναι τελικά θετική για το ευρώ και για τις χώρες εκτός του ευρώ και φυσικά βρίσκεται στο συμφέρον τη ενιαίας αγορά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καταρχάς, ευχαριστώ για τη γρήγορη εξέταση αυτής της νομοθετικής πρότασης. Ευχαριστώ τα μέλη της Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων, ιδίως την κυρία Χούμπνερ, αλλά και τους σκιώδεις εισηγητές από τις πολιτικές ομάδες για τον επικοδομητικό διάλογο που είχαμε για το φάκελο αυτό τις τελευταίες εβδομάδες και μήνες. Τώρα που επιτεύχθηκε η πολιτική συμφωνία για το Τούπακ, η πρόταση αυτή είναι το επόμενο βήμα που πρέπει να λάβουμε για να ενισχύσουμε τους μηχανισμούς σταθεροποίησης και να τους επικαιροποιήσουμε. Θα έπρεπε να αποφύγουμε τον κίνδυνο να στραφούμε, να περιοριστούμε στην Ευρωζώνη. Και αυτό είναι ο στόχος της πρώτας επιτροπής που αναθεωρεί τα, τον υφιστάμενο κανονισμό ισολογισμών ο υφιστάμενος ε, κανονισμός δημιουργήθηκε μετά την δημιουργία του EFSF, του ESM και του μόνιμου ESM. Επιπλέον ο κανονισμός αυτός δεν λαμβάνει υπόψη τις πρόσφατες ε, αλλαγές στην οικονομική διακυβέρνηση που έχουν στόχο την ενίσχυση του συντονισμού σε οικονομικό και δημοσιονομικό επίπεδο, την νομοθεσία ιδίω το Τούπακ κυρίω. Στο πλαίσιο αυτό, η νέα πρόταση της Επιτροπής ε, ε, χρησιμοποιεί τον υφιστάμενο κανονισμό, αλλά πηγαίνει περισσότερο, περαιτέρω, παρέχοντας τα κράτη που δεν έχουν νόμισμα το ευρώ και άλλα οικονομικά εργαλεία, όπως ε, τους το, την πιστοτική γραμμή ενισχυμένων ε, παροχών ή την προληπτική γραμμή εξασφαλίζοντας ισότιμο πεδίο λειτουργίας και στις δύο κατηγορίες χωρών που έχουν το ευρώ νόμισμα και που δεν έχουν. Η... Απαιτείται να προχωρήσει γρήγορα ο κανονισμός αυτός γιατί η κρίση δεν περιορίζεται στις χώρες της Ευρωζώνης μόνο. Αντίστοιχη και αντίστοιχα εργαλεία χρηματοοικονομικής βοήθειας και εργαλεία διακυβέρνησης θα πρέπει να παρέχονται όπως και η σχετική νομοθεσία στα κράτη-μέλη της Ένωσης που δεν είναι στο ευρώ για να μην χρειαστεί τα κράτη αυτά να αντιμετωπίζουν την κρίση με τα χέρια δεμένα πίσω από την πλάτη τους. Χρειάζεται λοιπόν γρήγορη δράση που θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Οι ομιλητέ τώρα εξ ονόματος των πολιτικών ομάδων. Ξεκινάμε από το ΕΛΚ με τον κύριο Μάρκους Φέρμπερ. Δύο λεπτά. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι. Θα ήθελα καταρχήν να ευχαριστήσω ιδιαίτερα την εισηγητριά μας την κυρία Ντανίτα Χίμπνερ για μια εξαιρετική έκθεση την οποία μας έχει παρουσιάσει όπου έθεσε τον δάκτυλο επί των τύπων των ύλων. Ακριβώς ε, κατέδειξε τα προβλήματα τα οποία μπορεί να προκύψουν γιατί κάνουμε ρυθμίσεις για το, τα χρηματοπιστωτικά θέματα αλλά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απουσιάζει σε πολύ μεγάλο βαθμό από αυτή τη διαδικασία. Αυτή η ενδιάμεση έκθεση δυστυχώς αντιμετωπίζει τα κενά έδρανα του Συμβουλίου και ίσως η Κομισιόν θα πρέπει να αναλάβει το, να μεταφέρει στο Συμβούλιο τις αιτήσει, τα αιτήματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ώστε να ξέρει τελικά και το Συμβούλιο περί τίνος πρόκειται. Για τους Γερμανούς στο ΕΛΚ, εμείς έχουμε κάποιες ανησυχίες, κάποιες αμφιβολίες για τα θέματα αυτά, ιδίως σε ό,τι αφορά την ανακεφαλοποίηση των τραπεζών, τίθεται το θέμα της μεταρρύθμισης της συνθήκης για τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητος που παίρνει μια διαφορετική μορφή πλέον και ιδίως το θέμα της ε, μεταφοράς των μη χρησιμοποιημένων μέσων του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας ο οποίος θα εκπνεύσει εν καιρό καταλήγουμε τώρα σε μια ανάμειξη μεταξύ χωρών που ανήκουν στη ζώνη του ευρώ και αυτών που δεν ανοίγουν στη ζώνη του ευρώ Πιστεύουμε ότι γενικά κινείται αυτή η έκθεση προς τη σωστή κατεύθυνση. Το ΕΛΚ θα την υποστηρίξει, αλλά έχουμε πολλές ανησυχίες από την πλευρά του, της Τσεντεού Τσέσου. Ευχαριστώ. Ακολουθεί ο κ. Κούτας από τη Σοσιαλιστική Ομάδα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Πίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι, πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Χίμπνερ για την εξαιρετική συνεργασία που είχαμε ήταν ε, απόλυτα διατεθειμένη να λάβει υπόψη και τις δικές μας προτάσεις ε, στις ε, συμβιβαστικές αυτής της έκθεσης. Τώρα, προτινόμενος κανονισμός για αυτό τον μηχανισμό χρηματοοικονομικής συνδρομής προς τα κράτη-μέλη που δεν έχουν ενταχθεί στην Ευρωζώνη έρχεται να διασφαλίσει ίσους όρους λειτουργία και ανταγωνισμού αν θέλετε σε μια περίοδο που η οικονομική κρίση έχει επηρεάσει όλα τα κράτη-μέλη σε ό,τι αφορά την αύξηση του δημοσίου χρέου και το καθεξής. Τώρα, έχουμε τις ε, χώρε τη Ευρωζώνης που έχουν αυτόν τον Ευρωπαϊκό ε, Μηχανισμό Σταθερότητας με τα 500 ε, δις ευρώ. Όμως, από την άλλη, τα κράτη-μέλη που δεν ανήκουν στην Ευρωζώνη έχουν μόλις 50 δις. Από τα 12 πήγαμε στα 50 βέβαια, όμως ο συνολικός αριθμός είναι κατά πολύ μικρότερο ε, του ποσού που έχουν στη διάθεσή του ε, τα κράτη-μέλη της Ευρωζώνη. Η Επιτροπή θέλει να θεσπίσει παρόμοιε διαδικασίε για ε, δάνεια παρόμοια με αυτά που ε, λαμβάνουν ε, τα κράτη-μέλη της Ευρωζώνης. Γι' αυτό στηρίζω την ιδέα αυτή της ε, ε, θέσπισης και εισαγωγή μηχανισμών ανακεφαλοποίησης τραπεζών για τα κράτη-μέλη εκτός Ευρωζώνης. Αυτές οι χώρες χρειάζονται έναν μηχανισμό τέτοιας προστασίας. Βέβαια θα ήταν καλύτερο να έχουμε έναν, έναν μηχανισμό άμεσης ανακεφαλαιοποίηση για να μην υπάρχει διαχωρισμός στην αγορά και έλλειψη ανταγωνιστικότητας. Eh, ευχαριστώ πρόεδρε και ευχαριστώ την κυρία Χιούμπνερ. Εξαιρετική δουλειά. Κατάφερε να λάβει την υποστήριξη όλων. Στην περίοδο αυτή οικονομικής κρίσης η Ένωση πρέπει να μείνει ενωμένη από το Βορρά και το Νότο. Αυτό είναι το πιο σημαντικό νομίζω και το έφηξε και ο Επίτροπος Ίσως οι χώρες εκτός της Ευρωζώνης να χρειάζονται υποστήριξη κατά τη διάρκεια της κρίσης και πρέπει να δημιουργήσουμε τις δυνατότητες ε, που να παρέχουν αυτή την ε, υποστήριξη. Χρειάζεται ξεχωριστό εργαλείο προφανώς από την Ευρωζώνη και έπρεπε να γίνει, αλλά πρέπει να αναθεωρήσουμε τώρα τα εργαλεία που έχουν στη διασύνη τους οι χώρες εκτός Ευρωζώνης. Με αυτό το κείμενο αυτό θέλουμε να πετύχουμε. Θα μπορούσαμε ωστόσο να προχωρήσουμε παραπέρα. Ακού, άκουσα βέβαια τον κύριο Φέρμπερ που είναι μια θέση που συμμερίζονται και κάποιοι στην ομάδα μου ότι αν ανοίξουμε το δρόμο σε νέα δημοσιονομικά εργαλεία θα πρέπει να αποφύγουμε να μπαίνουν ε, από την πίσω πόρτα του στο SSM ή το ESM. Αλλά δεν είναι αυτό το θέμα. Μετά από μακρά συζήτηση προσθέσαμε, προσφέραμε μια προσθήκη που, στο κείμενο που νομίζω θα αποδεχθεί η κυρία Χούμπνερ και που ελπίζουμε στην παράγραφο 7 ιδίω να γίνει δεκτή. Εμείς λέμε υπό τους όρους ε, συμμετοχής, ε, μόνιμης ε, συμμετοχής στο ESM και στο SSM και παρέχει τις ίδιες υποχρεώσεις και δικαιώματα όπως τα κράτη-μέλη. Αυτό είναι μια συμβιβαστική λύση για να μπορέσει η ομάδα μου συνολικά να υποστηρίξει την πρόταση της κυρίας Χιούμπνερ. Ευχαριστούμε εκ μέρους του ECR, ο κύριος Ζήλε. Es arī gribētu sākt ar pateicību <clears throat> par šo ziņojumu, lai arī, kā mēs zinām un dzirdam, te būs daudz pretrunīgu viedokļu. Θέλω να συνεχίσω εκεί που σταμάτησε η κυρία Νταρίτα Χίπνερ. Αυτή η έκθεση είναι μια προσπάθεια στα πλαίσια της κρίσης να υπάρξει ένα μηχανισ... ένας μηχανισμός προσανατολισμού και υποστήριξης για χώρες που δεν είναι μέλη της ζώνης του ευρώ με διευκολύνσεις όπως η προληπτική χρηματοδότηση και άλλες. Αυτό είναι πάρα πολύ θετικό. Οι χώρες οι οποίες θα ε, μπουν στο μηχανισμό εποπτείας θα μπορούν να έχουν τα, την ε, υποστήριξη για αυτόν τον μηχανισμό χωρίς να είναι ακόμα μέλη του, της ζώνης του ευρώ τα 10 δισεκατομμύρια τα οποία θα μεταφερθούν από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθεροποίησης θα περάσουν σε αυτή τη διευκόλυνση για το ισοζύγιο πληρωμών. Εδώ υπάρχουν ενδεχομένω ε, απόψεις ε, αρνητικές από ορισμένε χώρες που είναι δωρητές για αυτό το μηχανισμό. Ε, υπάρχουν αμφιβολίες γιατί κάποιες χώρες μπορούν να επιλέξουν να μπουν σε αυτό το μηχανισμό χωρίς να αποδεχθούν το ενίο καθεστώς ε, για την τραπεζική επίλυση. Για το λόγο αυτό η ομάδα μας έχει προτείνει μια σειρά από χωριστές ψηφοφορίες. Εγώ θα υποστηρίξω την έκθεση, άλλοι συνάδελφοι της ομάδας μας θα στραφούν εναντίον. <clears throat> Ελπίζω όμως, όπως είπε και ο κύριος Φέρμπερ, πιστεύω ότι αυτή η έκθεση δεν θα απορριφθεί παρόλα αυτά. Ο κύριος Χουντής, επόμενος μιλητής. Αγαπητοί συνάδελφοι, για δύο βασικούς λόγους η ομάδα μου δεν θα υποστηρίξει την έκθεση της κυρίας Χούμπνερ. Ο πρώτος είναι ε, ότι η έκθεση αναφέρεται βεβαίως σε μια προσπάθεια της Κομισιόν για να επικαιροποιήσει τον κανονισμό για το μηχανισμό ισοζυγίου πληρωμών για τα κράτη που δεν έχουν ως νόμισμα το ευρώ. Πρώτο πρόβλημα. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε αυτή τη διαδικασία δεν έχει τη δυνατότητα να παρέμβει επί της ουσίας, δεν έχει τη δυνατότητα να καταθέσει τροπολογίες επομένω η σύνταξη τη έκθεση το αναγνωρίζει ε, αν δεν κάνω λάθο και η συγγήτρια είναι επικουρική είναι συμβολική είναι για να κρατηθούν τα προσχήματα τη δημοκρατική νομιμοποίηση. τίθεται αγαπητοί συνάδελφοι για άλλη μια φορά το θέμα το πώ λαμβάνει αποφάσει και υιοθετεί κανονισμού η κομισιόν και πώ περιορίζεται ο ρόλο του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου. και ο δεύτερο λόγο αγαπητοί συνάδελφοι είναι το γεγονό ότι τόσο η πρόταση τη ε, κομισιόν όσο και η έκθεση υιοθετεί ότι τα μέτρα αυτά αυτό ο μηχανισμό, αυτή η υποστήριξη αυτά τα εργαλεία χρησιμοποιούνται για να υπάρχει ισότιμη μεταχείριση μεταξύ των χωρών εντό του ευρώ και εκτό του ευρώ. κατά τη γνώμη μα, αυτό είναι ένα προσχηματικό επιχείρημα διότι ουσιαστικά πρόκειται για μια οργανωμένη προσπάθεια τη κομισιόν να περάσει του μονοδρόμους τους νεοφιλελεύθερους μονοδρόμους της ύφεσης και τη λιτότητα και στι χώρε που είναι εκτό ευρώ τη συνταγή την ξέρουμε την έχουμε ζήσει στις χώρες εντός του ευρώ στην ελλάδα στην πορτογαλία και ούτω καθεξής. επομένως μια ισότητα που εξασφαλίζεται στη βάση βαθύτερης ύφεσης λιτότητας φτώχειας και ανεργίας δεν μας βρίσκει σύμφωνος. για αυτούς τους λόγους θα καταψηφίσουμε την έκθεση. ευχαριστώ πολύ κύριε πρόεδρε. πολύ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Να δώσω συγχαρητήρια στην κυρία Χιούμπνερ, η οποία έκανε ένα εξαιρετικό έργο στη συγγήτρια. Στις χώρες της ζώνης του ευρώ, στις ζώνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπάρχουν οι χώρες που δεν είναι μέλη της ζώνης του ευρώ και οι χώρες αυτές επλήγησαν και αυτές από την ε, κρίση και έχουν χωριστεί σε δύο ομάδες. Το γεγονός ότι έχουμε Τώρα, αυτή τη διάσπαση μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση μας οδηγεί σε αμφιβολίες για το αν μπορούμε πράγματι να λειτουργήσουμε σαν μια ενιαία οντότητα. Είναι απαραίτητο να γεφυρώσουμε το χάσμα μεταξύ των δύο αυτών ομάδων χωρών και αυτός είναι και ο στόχος αυτής της πρότασης που θέλει να διευκολύνει και τη λειτουργία του μηχανισμού υποστήριξης του ισοζυγίου πληρωμών. Με τον τρόπο αυτό θα είναι πιο εύκολο να ξεπεριστούν τα προβλήματα. Αλλά χρειαζόμαστε και περαιτέρω συστατικά στοιχεία για να εξασφαλίσουμε τη σταθεροποίηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Είναι απαραίτητο να εξασφαλίσουμε και την αλληλεγγύη αλλά και την βιωσιμότητα των μέτρων αυτών. Είναι σαφές ότι για να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε αυτή την κρίση θα πρέπει να υπάρξει και μεγαλύτερη πειθαρχία στον προϋπολογισμό και στο ισοζύγιο πληρωμών και αυτό επομένως θα πρέπει να καταγραφεί και σε συνταγματικό επίπεδο στις χώρες αυτές. Επίσης θα πρέπει να εξασφαλίσουμε το ότι ακόμα και στις χώρες αυτές που δεν είναι μέσα στη ζώνη του ευρώ μπορεί να υπάρξει ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών και με τον τρόπο αυτό μπορούν να τεθούν τα δημόσια οικονομικά σε βιώσιμη βάση με την μη περαιτέρω διόγκωση του κρατικού χρέους. Και έτσι μπορούμε να εξασφαλίσουμε ότι θα κινηθούμε προς την κατεύθυνση της εξυγένσης ακόμα και των χωρών αυτών που δεν είναι μέσα στη ζώνη του ευρώ. Βέβαια δεν μπορούν να επιληθούν αυτή τη στιγμή όλα τα λεπτομεριακά προβλήματα σε αυτή την έκθεση, αλλά πιστεύω ότι η τελική μορφή του κανονισμού θα πρέπει να τα αντιμετωπίσει όλα αυτά. Και εμείς θα υποστηρίξουμε φυσικά. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εγώ είμαι απόλυτα σύμφωνο με την έκθεση της κυρία Τανούτα, διότι και η χώρα μου που δεν είναι μέλος τη ζώνη του ευρώ, η Ουγγαρία, θα πρέπει και αυτή να τύχει μια υποστήριξη, όπως και οι χώρες της ζώνης του ευρώ. Εάν λοιπόν η Ουγγαρία, η Πολωνία, η Τσεχική Δημοκρατία αντιμετωπίσουν προβλήματα με τις τράπεζές τους και αυτές οι τράπεζες των χωρών αυτών φυσικά μπορούν να έχουν θηγατρικές σε χώρες της ζώνης του ευρώ, τότε μπορούν και αυτές οι τράπεζες να υποστηριχθούν. Κατανοώ λοιπόν αυτά τα οποία λέει η κυρία Χίμπνερ. Και επίσης θέλω να τονίσω ότι αν δεν υπάρξει ίση μεταχείριση όλων των τραπεζών στην Ευρώπη, ίση μεταχείριση όλων των τραπεζικών λογαριασμών, αυτό μπορεί να οδηγήσει σε μια κατάσταση όπου θα διασπαστεί και θα κατακαιρματιστεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, τουλάχιστον στη ζώνη του ευρώ και στους, στις χώρες που είναι εκτός της ζώνης του ευρώ. Αυτό θα είναι λάθος για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο κύριος Γκούσταυσον. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εκτός ε, του Κοινοβουλίου καταλύονται όλοι οι μηχανισμοί πρόνοιας από τα μέτρα οι πολίτες μας οδηγούνται στη φτώχεια και όλα αυτά λόγω ε, της περιορισμένης, ε, του περιορισμένης θεώρησης ε, της Τρόικας που δεν βλέπει το σύνολο της οικονομίας, έχει μια αποσπασματική θεώρηση. Πολλοί από εμάς θέλουμε μια αλλαγή, θέλουμε να βάλουμε τους ανθρώπους μπροστά από τα κέρδη και τα χρήματα. Όμως ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση ακολουθεί πάντα τους δικούς μας ε, στόχους και έτσι έχουμε τα παλιά και γνωστά. Η κυρία Βίμπνερ προτείνει μια επανάληψη με, με τα όσα των όσων ισχύουν για τις χώρες ε, της Ευρωζώνης. Ε, αν όμως και εκεί υπάρξουν οικονομικά προβλήματα, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα τις ε, κατακλείσει με τέτοιες νεοφιλελεύθερες πολιτικές. Όμως στο τέλος καταλήγουμε σε αρνητικές συνέπειες. Υπάρχει ένα ερώτημα προς εσάς από τον κύριο Σμιτ. Θέλετε να το απαντήσετε? Κύριε Σμιτ. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Γούσταυσον πού ακριβώς στην έκθεση της κυρίας Χούμπνερ ε, είχατε, ε, βρήκατε αυτό τον πονόκυλο ε, στον οποίο ενδεχομένω να παραπέμπετε. Προσπαθήσατε να συνοψίσετε το κείμενο, νομίζω ότι δεν το κάνατε σωστά. Το Λάθο το είπατε. Ακριβώς ε, με την επίλυση των κρίσεων. Ε, για αυτό το ζήτημα μιλάμε. Και πρέπει να γίνεται με τους ίδιους όρου και με τις ίδιες συνθήκες που γίνεται παντού. Αυτό κάναμε και στη δεκαετία των 90 που υπάρχει αυτή η παραπομπή ε, στον πονόκυλο που λέτε ο κύριος Σμιτ πού ακριβώς βρισκόταν τα τελευταία πέντε χρόνια όταν είχαμε όλες αυτές τις πολιτικές. Δεν ήσασταν εδώ προφανώς. Είναι η ίδια αυτή η πολιτική. Αν δείτε αυτά τα ε, μακροοικονομικά μέτρα που ε, εφαρμόζονται παντού με τους ίδιους κανόνες για τις νέες χώρες, θεωρείται δίκαιο και αυτέ οι χώρε και αυτέ που δεν βρίσκονται στην Ευρωζώνη να έχουν του ίδιου όρου. σω να είναι δίκαιο, αλλά είναι οι ίδιε πολιτικέ λιτότητα. Δεν θα πάρουν μέτρα αν δεν κάνουν ακριβώ τα ίδια με τι υπόλοιπε χώρε, δηλαδή να περικοπές μισθών, συντάξεων και το καθεξής. Ευχαριστώ. Ε, κυρία Κλέβα Τα τελευταία δύο χρόνια στην Ευρώπη εισήχθησαν πολλά νέα εργαλεία χρηματοοικονομικής βοήθειας στην Ευρωζώνη, απαντώντας στις πιέσεις και τις επιπτώσεις της οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσεως. Το EFSF, ιδρύθηκε το EFSF, ε, εγκρίθηκε το ESM, για να αντιμετωπίσουν την κρίση του ευρώ. Η κρίση ωστόσο και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν ορισμένα κράτη της Ευρωζώνης κατέστησε σαφές ότι η Ευρώπη πρέπει να ορίσει έναν ειδικό μηχανισμό που θα μπορούσε να αποφύγει την διάδοση του προβλήματος. Αυτή ήταν η πρόταση λεγόμενη BOP που μπορεί να βοηθήσει και τις χώρες, τις χώρες εκτός Ευρωζώνης πρόοδος που πετύχαμε με το πρόσφατο Τούπακ και οι νέες διατάξεις ε, της ΕΡΚ ΕΕ που περιλαμβάνονται στην έκθεση Φεραίρο πρέπει να ενισχυθούν με νέα χρηματοπιστωτικά εργαλεία προς τα κράτη που δεν έχουν το ευρώ ως νόμισμά τους. Καλωσορίζω την συμπερίληψη της ανάγκης να υπάρχει ε, μελέτη κόστου ως όφελος για τις δημόσιες επενδύσεις και την, ενώ η, το εργαλείο αυτό για τις χώρες εκτός ε, ευρώ θα πρέπει να προβλέπουν έλεγχο των δημοσίων οικονομικών καθώς και προβλέψεις για τις επιπτώσεις που θα έχουν συγκεκριμένα δημοσιονομικά μέτρα για την Ευρώπη του 2020. Ο κύριος... Δύο λεπτά για τον κύριο Στόλογιαν. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρο. Η χώρα μου, η Ρουμανία, έχει πάρει χρηματοδοτική υποστήριξη από την Ευρωπαϊκή Ένωση σε μια πολύ δύσκολη χρονική στιγμή μέσα στην κρίση. Θα ήθελα εδώ να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου σε όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα για το γεγονός αυτό. Αλλά όταν βρίσκεται σε δυσκολία μια χώρα που δεν είναι στη ζώνη του ευρώ, έχει την εντύπωση ότι δεν την χάνουν τις ίδιες μεταχείρισεις και δεν έχουν την ίδια πρόσβαση στο οπλοστάσιο μέτρων χρηματοδοτικής υποστήριξης όπως οι χώρες του ευρώ. Για το λόγο αυτό θέλω να υποστηρίξω απόλυτα την πρόταση της κυρίας Χίπνου, της εισηγητριάς μας, για να μπορέσουμε <clears throat> να θίξουμε αυτό το θέμα. Και υποστηρίζω ιδιαίτερα την πρόταση να υπάρξει αυτό το ιδιαίτερο χρηματοδοτικό εργαλείο για την ανακεφαλαίωση τραπεζών χωρών που δεν βρίσκονται στη ζώνη του ευρώ. Θα πρέπει να υπάρξει φυσικά αιρεσιμότητα μέσα στα πλαίσια αυτά για υγιείς οικονομικές και χρηματοπιστωτικές πολιτικές. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Οντί έχει το λόγο τώρα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε και εγώ θα ήθελα να συνταχθώ με όλους αυτούς που επίνεσαν την κυρία Ντανίτα Χίμπνερ και επίση να ευχαριστήσω εσά, κύριε Επίτροπο για την προσπάθεια που είτε κάνει να εξασφαλιστεί τη σταθερότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο αφορά το μηχανισμό χρηματοδοτική υποστήριξη σε περίπτωση απειλών για το ισοζύγιο πληρωμών χωρών που το νόμισμά του δεν είναι το ευρώ, με νομική βάση το άρθρο 143 τη συνθήκη. Και εδώ υπάρχει ένα όριο 50 εκατομμυρίων, αλλά με την επιφύλαξη μακροοικονομικής προσαρμογής και εποπτείας σε ό,τι αφορά την εφαρμογή των μέτρων αυτών. Όπως είπατε κύριε Πρόεδρε, η νέα πρόταση τώρα αντικαθιστά το ευρωπαϊκό εξάμεινο και τη διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος με την τροποποίηση του προηγούμενου κανονισμού. Αλλά Θέλω να θέσω το εξή ερώτημα. Για τι χώρε τη ζώνη του ευρώ έχουμε την διεθνή αυτή συμφωνία, τη διακρατική συμφωνία που είναι ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθεροποίηση. Αναφερθήκατε σε όλα τα εργαλεία τα οποία συνηγορούν υπέρ τη προτάσεω σα, Αλλά όλα αυτά είναι μηχανισμοί οι οποίοι θα πάψουν να υπάρχουν όπως το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και ο Μηχανισμός Σταθερότητας, το ESM. Γιατί λοιπόν αυτή η νομική βάση να εδράζεται στο άρθρο 143. Δεύτερον, πώς συνδέονται όλα αυτά με το συντονισμό των οικονομικών πολιτικών και το σύμφωνο σταθερότητας. Υπάρχουν χώρες που έχουν την πλήρη επιλογή του opt-out από την ζώνη του ευρώ. Πώς συνδυάζεται αυτό με το σύμφωνο σταθερότητας και γιατί στο άρθρο 6 θέλετε να υποχρεώσετε τις χώρες να υφίστανται αυτή την αυξημένη επιτήρηση ενώ είναι κυρία κράτη. Ευχαριστούμε. Ένα λεπτό για τον κύριο Βάλτσιτης. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για την πρόταση που έχει προετοιμάσει. Νομίζω ότι η αναθεώρηση του υφιστάμενου κανονισμού είναι επίκαιρη γιατί ε, οι χώρες εκτό Ευρωζώνης θα πρέπει να, έχουν, να λαμβάνουν χάγια για την ε, ανάληψη βοήθειας γιατί είναι δύσκολε οι οικονομικές συνθήκες. Όμως ε, αναφερθήκατε στην ανακεφαλοποίηση του τραπεζικού τομέα. Αυτό θα πρέπει να γίνεται ανοιχτά και σε ό,τι αφορά τη λειτουργία των τραπεζών. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το στοιχείο και, και υπό το φως της ε, κρίσης. Γι' αυτό σε όλα αυτά τα κείμενα θα πρέπει να μιλάμε για μεγαλύτερη υπευθυνότητα των ε, ε, τραπεζικών φορέων. Αν θέλουμε να επιλύσουμε το ζήτημα της χρεοκοπίας τραπεζών, τα κράτη-μέλη θα πρέπει να έχουν τους διορθωτικούς δείκτες Δηλαδή τα κράτη-μέλη θα πρέπει να καλύψουν ε, τις δαπάνες. Γι' αυτό ελπίζω οι νέες ε, διατάξεις και η πρόταση της Επιτροπής θα έχει μεγαλύτερη ε, ευθύνη του τραπεζικού τομέα. Περνάμε στη δικασία Catch the με πέντε μέλη που έχουν ζητήσει το λόγο. Ο κύριος Νικολάς. Ευχαριστώ. Επίτροπε συνάδελφοι, η παγκόσμια οικονομική κρίση είχε αντίκτυπο σε όλα τα κράτη της Ένωσης. Σήμερα δεν είμαστε ακόμα σε θέση να ξεπεράσουμε την ύφεση. Δεν πρέπει λοιπόν να διακρίνουμε μεταξύ χωρών της Ευρωζώνης και χωρών εκτός Ευρωζώνης. Όλοι στο ίδιο βαπόρι είμαστε. Πρέπει λοιπόν να προσέχουμε ε, μη τυχόν υπά, λάβουμε μέτρα που οδηγήσουν σε ακόμα μεγαλύτερη μακροοικονομική ανισορροπία. Βλέπουμε ότι δημιουργείται σιγά σιγά μια τραπεζική ένωση, ένα μελλοντικό σημαντικό εργαλείο αντιμετώπισης περίπλοκων χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Είναι σημαντικό τα μέλη της Τραπεζικής Ένωσης να έχουν επαρκείς ε, πόρους για να διατηρήσουν την σταθερότητα του νομίσματος. Για να μπορέσει η Τραπεζική Ένωση να λειτουργήσει θετικά για όλη την Ένωση θα πρέπει να υπάρχουν κονδύλια για την αντιμετώπιση των κλήσεων και να διατίθενται σε όλους. Επόμενος μιλητής. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Πιστεύω ότι η σταθερότητα είναι πολύ σημαντική για τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι χώρες που έχουν ελληματικό προϋπολογισμό ε, είναι αρκετές, αλλά στην ε, Ουγγαρία μένει κάτω από το 3% από το 2010 και έχει μειωθεί πράγματι το έλλειμμα. Η... Εκτός από την Ουγγαρία μόνο άλλα τέσσερα κράτη-μέλη έχουν επιτύχει κάτι τέτοιο. Δεν έχει ζητήσει η Ουγγαρία λοιπόν βοήθεια Παρά το γεγονό ότι το 2010 βρεθήκαμε σε πολύ πιο δύσκολη κατάσταση από την Ελλάδα. Η διαχείριση κρίση τη ουγγρική κυβέρνηση ήταν υποδειγματική. Και ένα παράδειγμα για τι άλλε χώρε Ευρωπαϊκή Ένωση. Για μα είναι όμω απαραίτητο ακόμα και οι χώρε που δεν είναι στη ζώνη του ευρώ να πάρουν μια <clears throat> υποστήριξη όπω ακριβώ και οι χώρε οι οποίε ανήκουν στη ζώνη του ευρώ. Ακολουθεί ο κ. Πάσκο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Είναι φυσικό ότι όπως και οι χώρες της Ευρωζώνης και οι υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορούν να χρειαστούν βοήθεια για να ανακεφαλαιώσουν τις τάπεζές τους. Ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας έχει δημιουργηθεί για να αντιμετωπίσει κινδύνους στη ζώνη του ευρώ και στην τωρινή της μορφή, τωρινή του μορφή δεν είναι έτοιμο για να αντιμετωπίσει τα προβλήματα χωρών εκτό τη ζώνη του ευρώ. Η έκθεση τη κυρία Φίμπνερ παρουσιάζει δύο επιλογέ για το πώ να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών σε χώρε που δεν είναι μέλη τη ζώνη του ευρώ. Από την έποψη της νομικής ασφάλειας πιστεύω ότι είναι πολύ καλύτερο να ακολουθήσουμε την επιλογή αυτή που ζητά την αλλαγή της συνθήκης για την δημιουργία του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας ότι τα κράτη-μέλη μπορούν να συμβάλλουν για το κεφάλαιο του φορέα αυτού που εξασφαλίζει την δυνατότητα διάσωσης και ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών. Η άλλη επιλογή <clears throat> η οποία αναφέρεται, παροχή δηλαδή δανείων για τις χώρες εκτός του, της χώρας του ευρώ, αυτό νομίζω ότι μονάχα θα παγίωνε τις διαφορές μεταξύ των χωρών της Ευρωζώνης και των χωρών μη στην Ευρωζώνη. Η κυρία Μπασέσκου. Ευχαριστώ. Η αναθεώρηση του υφιστάμενου οικονομισμού μπορεί να επιτρέψει σε κράτη-μέλη που δεν έχουν το ευρώ να αποκτήσουν εργαλεία παρόμοια με τα όσα έχουν οι χώρε τη Ευρωζώνη. Η χώρα μου ήταν μία από τι πρώτε που επωφελήθηκαν οικονομική στήριξη από την Ευρωπαϊκή Ένωση χάρη στον μηχανισμό, ε, μηχανισμό συνδρομής ε, BOP του ισολογισμού. Ε, ενώ καταφέραμε να σταθεροποιήσουμε τα δημοσιοοικονομικά μας ε, και να ξεκινήσουμε μια σειρά σημαντικών μεταρρυθμίσεων. Όμως ε, το πολιτικό κόστος ήταν εξαιρετικά υψηλό. Καταφέραμε όμως να μειώσουμε το δημοσιονομικό μα έλλειμμα και να θέσουμε από έλεγχο το χρέος. Όμως τώρα υπάρχει ο κίνδυνος δεσμεύσει στην υφιστάμενη συμφωνία με την Επιτροπή και το Γεθνή Νομισματικό ταμείο να μην ε, εκπληρωθούν από τη σοσιαλιστική κυβέρνηση. Έτσι μπορεί να τεθεί ε, εν αμφιβόλο όλες οι προσπάθειες ε, μεταρρύθμισης που έχουν καταβάλει προηγούμενες κυβερνήσεις. Ευχαριστούμε. Ο κ. Λουχάν. Ευχαριστώ. Η οικονομική κατάσταση των τελευταίων ετών δημιούργησε σημαντική οικονομική βλάβη στην οικονομία αύξησε τα ελλείμματα και δημιούργησε σοβαρά προβλήματα εντός και εκτός Ευρωζώνης. Ε, τα κράτη η κρίση μπορεί να περάσει και στα κράτη που είναι εκτός ευρώ, στα κράτη της Ένωσης που είναι εκτός ευρώ, εύκολα. Γι' αυτό πιστεύω ότι οι χώρες που μετέχουν στον ενιαίο μηχανισμό εποπτείας θα έπρεπε να μετέχουν και στο ESM και ιδίω δε στο εργαλείο ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών. Οι περισσότερε χώρες ε, δυσκολεύονται να έχουν πρόσβαση στα ενωσιακά χρηματοοικονομικά εργαλεία. Η αύξηση λοιπόν της χρηματοδότησης, της χρηματικής βοήθειας μέσω της ε, διαδικασίας αυτής θα αυξήσει και την δυνατότητα απορρόφησης των πόρων από τις χώρες αυτές. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Η οικονομική κρίση επηρέασε σημαντικά τους προϋπολογισμούς των κρατών. Τούτο οδήγησε σε αύξηση των πόρων, στα 50, των διαθέσιμων πόρων στα 50 δις. Δόθηκαν, διατέθηκαν σημαντικά ποσά στι χώρε που αντιμετωπίζουν δυσκολίε, μεταξύ των οποίων και τη χώρα μου, τη Ρουμανία. Ωστόσο, παραμένει προβληματική υλοποίηση του μηχανισμού, διότι τα κράτη-μέλη τη Ένωση που δεν είναι μέλη του ευρώ δεν έχουν πρόσβαση στα ίδια χρηματοοικονομικά εργαλεία όπω και οι χώρε τη Ευρωζώνη. Πρέπει να υπάρχει ισότιμη ε, πεδίο ε, συγκρίσιμη δυνατότητα στον τομέα αυτό το οποίο δεν, δεν πραγματοποιείται αυτή τη στιγμή. Ε, η κατάσταση ό,τι αφορά το ισοζύγιο πληρωμών και τους BOP μπορεί να διευκολύνουν ε, την απορρόφηση ευρωπαϊκών πόρων και την αντιμετώπιση της κρίσης. Υποστηρίζω απόλυτα την έκθεση Χούμπνερ και τη συγχαίρω για την εξαιρετική έκθεσή της. Ευχαριστώ πολύ και τώρα κλείνουμε τη συζήτηση. Θα δώσω καταρχήν το λόγο στον κύριο Ρεν, εξ Κομισιόν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, έντιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την πάρα πολύ ουσιαστική συζήτηση που έχει γίνει για αυτό το τόσο σημαντικό θέμα για την Ευρωπαϊκή Ένωση στο σύνολό της και ολόψυχα υποστηρίζω την ε, έμφαση που έθεσε η κυρία Χιούμπνερ στην ανάγκη να διατηρηθεί η συνοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό αναφέρθηκε και από πολλούς ε, ομιλητές στη σημαίνει συζήτηση. Ακόμα δεν γνωρίζουμε ποια θα είναι τα σημαντικά θέματα τα οποία θα αντιμετωπιστούν από το Συμβούλιο, γιατί δεν έχει ακόμα ξεκινήσει τη διαπραγμάτευση εκεί. Γι' αυτό η θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι πάρα πολύ καλόδεκτη, γιατί θα βοηθήσει να εμπλουτίσει περισσότερο τις συζητήσεις στους κόλπους του Συμβουλίου. Θέλω να αδράξω αυτή την ευκαιρία για να ενθαρρύνω το Συμβούλιο να ξεκινήσει το ταχύτερο δυνατόν την επεξεργασία αυτού του θέματος. Θέλω επίση να ευχαριστήσω τον κύριο Στολογιάν και τον κύριο Οντί για το γεγονός ότι αναφέρθηκαν στις εμπειρίες της Ρουμανίας και στο θετικό αντίκτυπο του μέσου υποστήριξης του ισοζυγίου πληρωμών και την σταθερότητα, σταθεροποίηση και ανάκαμψη της Ρουμανίας. Τα τελευταία χρόνια και η Ουγγαρία και η Λετωνία έχουν επωφεληθεί από προγράμματα στήριξης του ισοζυγίου πληρωμών. Η εμπειρία της Λετωνίας είναι ιδιαίτερα εύγλωτη όταν η κρίση έπληξε την Ευρώπη ε, εισαγόμενη από τις Ηνωμένες Πολιτείες, έπληξε και την Λετωνία ιδιαίτερα η Λετωνία όμως υποστηρίχθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Μηχανισμού Στήριξης Ισοζυγίου Πληρωμών, του BOP. Επίσης υποστηρίχθηκε και από τις σκανδιναβικές χώρες και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Η Λετωνία εφήρμοσε ένα τολμηρό και απαιτητικό πρόγραμμα οικονομικών μεταρρυθμίσεων και δημοσιονομικής προσαρμογής και τώρα έχει ανακάμψει έχει βγει από το πρόγραμμα αυτό προσαρμογής, η οικονομία της ενισχύεται συνεχώς και βλέπουμε πολύ καλύτερες προς προοπτικές απασχόλησης στη Λετωνία. Δεν λέω ότι δεν θα προκύψουν δυσκολίες. Υπάρχουν δυσκολίες. Εξακολουθεί να είναι πολύ δύσκολο αυτό το πρόγραμμα προσαρμογής, αλλά είναι σαφές ότι η Λετωνία έχει περάσει ένα σημαντικό σκόπελο και μπορεί να προχωρήσει με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σήμερα η Λετωνία είναι ένας ε, σοβαρός υποψήφιος για να γίνει μέλος της ζώνης του ευρώ μετά από την Εστονία. Τώρα, σε σχέση με το θέμα της νομικής βάσης που ανέφερε ο κύριος Χουντής, η πρόταση αυτή βασίζεται στο άρθρο της συνθήκης. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί η διαδικασία σύμφωνη γνώμη από την πλευρά του Κοινοβουλίου. Ο κύριο Σοντή έθεσε και αυτό εύστοχα ερωτήματα. Μπορώ να σα υποσχεθώ ότι η Κομισιόν θα μπορέσει να σας δώσει πιο λεπτομερείς απαντήσεις σε αυτά τα σημαντικά ερωτήματα για να διευκρινιστεί το περιεχόμενο των προτάσεων αυτών. Συνεχίζω στα Σουηδικά για να απαντήσω στον κύριο Γκούσταυσον στην... Ε, και αναφέρομαι και στον κύριο Γούστασον και στον κύριο Σμίτ, οι οποίοι φυσικά μίλησαν και αυτοί ειδικά σήμερα. Θέλω απλώς να πω ότι η αλληλεγγύοι που επέδειξαν οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω μηχανισμών όπως αυτός που εξετάζουμε σήμερα θα εξασφαλίσουν και υποστήριξη για τις φτωχότερες χώρες και τους πληθυσμούς τους και μόνο με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να επιτύχουμε περαιτέρω ανάκαμψη και δημιουργία θέσεων απασχόληση, αφού προηγουμένω εξασφαλίσουμε την οικονομική σταθεροποίηση. Και αυτό είναι το αντικείμενο αυτή τη μετάρρυθμιση. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Επίτροπε. Και δίνω τώρα το λόγο στην κυρία Χιούμπνερ. Δύο λεπτά εισηγήτρια. Ευχαριστώ πολύ. Πολύ σύντομα θα ήθελα να απαντήσω σε δύο παρατηρήσεις από τον κύριο Φέρμπερ, συνάδελφο του ΕΛΚ, σε ό,τι αφορά τους προβληματισμούς του για την ανακεφαλοποίηση των τραπεζών και την πρόσβαση των χωρών εκτός Ευρωζώνης στην ανεκεφαλαιοποίηση τραπεζών και αντίστοιχου ταμείου. Να πω ότι το Κοινοβούλιο μα ε, σχετικά πρόσφατα υιοθέτησε το μηχανισμό του opt-in για τις χώρες εκτός Ευρωζώνης ε, ως προς τον ενιαίο εποπτικό μηχανισμό και ξέρουμε ότι σε αυτό το μηχανισμό ίσως να βρεθούμε σε περιπτώσεις όπου ο επόπτης θα θέσει ε, συστάσεις στον εθνικό χρηματοπιστωτικό τομέα ή ακόμα και περιποθέσεις ε, που θα, ενδεχομένως να οδηγήσουν σε ανακεφαλοποίηση των τραπεζών. Νομίζω λοιπόν ότι η ευθύνη μας θα πρέπει να υπερβαίνει τον ενιαίο εποπτικό μηχανισμό και να δούμε πώς μπορούμε να βοηθήσουμε και όλα ε, τα κράτη-μέλη αυτά για να έχουν πρόσβαση στην ανακεφαλοποίηση βάση δανείων, βάση δανεισμού. Δεύτερον, ε, όταν μιλάμε για την μεταφορά από το EFSM που θα σταματήσει σύντομα όταν θα τεθεί σε ισχύ ο ESM, η μεταφορά δεν αφορά την μεταφορά εναπομείναντων πόρων, αλλά δαν, δανειακής, ε, δανειακού δυναμικού, αν θέλετε, capacity. Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω όσους, όσοι συνεργάστηκαν μαζί μου ε, τους τελευταίους μήνες, τους εσκιώδεις και όσους συμμετείχαν σε αυτό τον εξαιρετικά πλούσιο διάλογο σήμερα. Ευχαριστούμε πολύ. Κλείνουμε λοιπόν αυτή τη συζήτηση. Η ψήφο θα λάβει χώρα αύριο στις 11.30 ψηφοφορία. Συγγνώμη. Παίρναμε τώρα στο επόμενο σημείο της ημερήσια διάταξης. Προφορική ερώτηση προ την Επιτροπή για τις ε, περιφερειακές κρατικές ενισχύσει. Bardzo proszę o zabranie głosu